Okay, colleagues, I think we should make a start because it's no. Ναι. time is pressing. The Commission's been waiting. So, um... Ε, συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε ε, με το σημείο 9 της Μέσης Διάταξης, όπου θα συζητήσουμε δύο σημαντικές ανακοίσεις από την πλευρά της ε, Επιτροπής τι οποίε λάβαμε την ε, προηγούμενη εβδομάδα και είναι πολύ σημαντικέ για την Επιτροπή μα. Η πρώτη από αυτέ είναι η εταιρική σχέση χωρών και Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μετά το 2020 και από εκεί και μετά η, η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και έχουμε μαζί τον Επίτροπο Μέμιτσα, ο οποίο θα μα παρουσιάσει αυτέ τι ανακοινώσει για τι χώρε ε, ΑΚΕ. Γνωρίζετε ότι έχουμε οθετήσει την έκθεση Νόιζερ Και Πράγματι υπάρχει, υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ της ανακοίνωσης και της έκθεσης γιατί χρειαζόμαστε νέα ε, στοιχεία και στο πλαίσιο της νέας κοινή αντίληψης. Και έχουμε προφανώς και το νέο ε, πλαίσιο, δηλαδή με το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο, την ατζέντα για το 2030 της βιώσιμης ανάπτυξης και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ευρύτερες αλλαγές ε, που λαμβάνουν χώρα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μογκερίνη την Τετάρτη στο Στρασβούργο, στη συνάντηση των συντονιστών, αναφέρθηκε στο στρατηγικό πλαίσιο εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρθηκε και στην ε, παγκόσμια στρατηγική. Οπότε έχουμε τα έγγραφά μα, έχουμε και τον εισηγητή μα εδώ, τον κύριο Νόιζορ. Οπότε σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σα σήμερα εδώ και σα δίνω το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε, συνάδελφοι, όπως πάντοτε αποτελεί τιμή και μένα το γεγονός ε, προσκαλείται εδώ για να μιλήσω στην Επιτροπή σας ε, και βέβαια έχουμε, ε, είχαμε πάντοτε μια στενή συνεργασία και σε σχέση με αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή την ανακοίνωση τόσο σε ό,τι αφορά την εταιρική σχέση με τις χώρες και όσο και σε ό,τι αφορά την ναι, νέα κοινή αντίληψη. Και η εργασίες μας ε, σε σχέση με αυτούς τους δύο φακέλους, με αυτά τα δύο ζητήματα έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, σε ένα ορόσημο και πραγματικά έχουμε σήμερα την πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε το τι θα γίνει από εδώ και στο εξή. Όπως γνωρίζετε την τελευταία εβδομάδα η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πακέτο προτάσεων ε, το οποίο περιλαμβάνει αυτές τις δύο ανακοινώσει. και υπήρξε και ένα τρίτο έγγραφο το οποίο ε, παρουσιάζει ένα ευρύτερο όραμα σε ό,τι αφορά ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό όραμα για την εφαρμογή της ε, ατζέντα του 2030, του θεματολογίου του 2030, τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε συνεργασία με τους εξωτερικούς μας εταίρους. Ε, διάβασα και το δικό σας σχέδιο έκθεση σε ό,τι αφορά τη νέα κοινή αντίληψη, που ε, δημοσιεύτηκε πριν από μερικέ μέρε. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου Νόιζερ και Δέγνα για αυτήν την έκθεση. Επίση, χαιρετίζω και ε, το πρόσφατο ψήφισμα πάλι από την πλευρά του κυρίου Νόιζερ ως εισηγητή ε, σε ό,τι αφορά ε, τις νέες σχέσεις, την νέα σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρων ΑΚΕ. Και βλέπω με ικανοποίηση ότι πραγματικά η σκέψη μας, η συλλογιστική μας μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου ευθυγραμμίζεται. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί ε, είχαμε τη δυνατότητα στο επίπεδο της Επιτροπής σας να ε, συζητήσουμε την ουσία των προτάσεών μας ε, και στη συνάντηση που είχαμε στα τέλη Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιο της συνάντηση των συντονιστών με την ύπατη εκπρόσωπο. θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει το περιθώριο για να δημιουργήσουμε μια κοινή βάση σε ό,τι αφορά τη σκέψη μας, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την νέα κοινή αντίληψη βλέπω στο δικό σας σχέδιο έκθεσης ότι η επίτευξη, η σύναψη μιας ε, συμφωνίας ε, σε συλλογική βάση αποτελεί προτεραιότητα τόσο για εσάς, για το Κοινοβούλιο, όσο και για εμάς την Επιτροπή. Και βλέπουμε ότι θεωρείται πως αυτή η κοινή αντίληψη έρχεται στο σωστό χρονικό ε, σημείο και είναι και απαραίτητη. Η Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει σε αυτό το πλαίσιο μια κοινή βάση για το κοινό μας όραμα, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στην ατζέντα του 2030 και προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες ε, προκλήσεις ενός όλο ένα και πιο παγκοσμιωμένου ε, και δικτυωμένου κόσμου. Και ε, σε αυτή τη στρατηγική θα πρέπει να ενταχθούν και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τα κράτη-μέλη. Και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι δηλαδή ω Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των SDGs ε, και να προσφέρουμε με αυτόν τον τρόπο ένα αντίβαρο ε, στην ρητορική του απομονωτισμού ε, η οποία βλέπουμε να κερδίζει σε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις κύριες κινητήρες δυνάμεις της ανάπτυξης ό,τι αφορά για παράδειγμα την ισότητα των φίλων, την νεολαία, την κλιματική αλλαγή, την ε, βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, θέματα τα οποία θίγει και η δική σας έκθεση. Και στον πυρήνα όλων αυτών βρίσκεται ο, βασικός μας στόχος, δηλαδή η εξάλληψη της ε, φτώχειας. Προτείνουμε λοιπόν τη δόμηση της ε, νέας κοινή αντίληψης πάνω σε αυτά τα, στις πέντε προτεραιότητες, δηλαδή άνθρωποι, πλανήτης, ευημερία, ειρήνη και εταιρική σχέση. Τα 5P όπως λέγονται. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο οι προτεραιότητες μας να είναι ορατές, να είναι ε, διασυνδεδεμένε μεταξύ τους ε, και σε αυτό το πλαίσιο η συνοχή της ε, πολιτικής στο επίπεδο της ανάπτυξης παίζει ένα πολύ κεντρικό ρόλο και βέβαια η δική σας Επιτροπή έχει αναφέρει με έμφαση την προτεραιότητα που έχει αυτή η διάσταση. Και η Επιτροπή σας έχει επίσης αναφέρει επανειλημμένα όλες τις διαστάσεις οι οποίες σχετίζονται ε, με τις δικές μας προτεραιότητες, δηλαδή ανθρωπιστική ε, βοήθεια, μεταναστευτική πολιτική, εμπορική πολιτική και άλλες. Και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα εφαρμογής και όλες τις εταιρικέ σχέσεις που έχουμε στη διάθεσή μας για να εφαρμόσουμε την κοινή αντίληψη. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει και να συμβάλλουν με το 0,7% του ακαθάριστο χώρο εισοδήματό του για την επίτευξη αυτών των στόχων και επίση ε, θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιτύχουμε του σχετικού ε, στόχου σε ό,τι αφορά τι ε, λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Επίση, οι εταιρικέ σχέσει με τι χώρε τη Μέση Ανατολή θα είναι πολύ σημαντικέ, ούτω ώστε να επιτύχουμε την ισότητα και μεταξύ των δύο φύλων και προκειμένου να προωθήσουμε και τα δημόσια αγαθά. Όπως σωστά αναφέρατε και εσεί, από την πλευρά του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε και ε, περαιτέρω μέσα χρηματοδότηση αυτών των στόχων, πέραν δηλαδή των ενισχύσεων, μέχρι για παράδειγμα μέσω κινητοποίησης των ε, δημοσίων κοντιλίων, αλλά και μέσω εταιρικών σχέσεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Οι προτάσεις μας για το Ευρωπαϊκό ε, Σχέδιο Εξωτερικών Επενδύσεων αποτελούν ακριβώς ένα παράδειγμα, αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής της νέας προσέγγισης ε, για την χρηματοδότηση που ακολουθούμε. Συμφωνώ επίσης μαζί σας ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα ε, της ανάπτυξης και όχι απλά να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προτείνουμε συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση μια πιο συντονισμένης προσέγγισης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών μέσω δηλαδή κοινών δράσεων, κοινών ε, προγραμμάτων και με λίγα λόγια θα πρέπει να καταφέρουμε περισσότερα, να καταφέρουμε καλύτερα τα όσα κάνουμε και να τα κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Ε, και τώρα να αναφερθώ στο ζήτημα των σχέσεων με τις ε, χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού. Από, διαφορετικές, από διάφορες απόψεις ουσιαστικά θα έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της νέας αυτής εταιρικής σχέσης και η ανακοίνωση της Επιτροπής ουσιαστικά αναφέρει τα βασικά ισχυρά σημεία και τα βασικά στοιχεία ε, πάνω στα οποία θα δομηθεί η νέα εταιρική σχέση. Βλέπω με χαρά μου ότι συμφωνούμε ως προς το ότι η συνεργασία μεταξύ ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο ε, που συνενώνει 110 ε, χώρες με 1,5 δις πολίτες σε ένα κοινό πλαίσιο αρχών. Αυτές οι κοινέ αρχές, δηλαδή η ειρήνη, η δημοκρατία, τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου, ε, παραμένουν όσοι έχουν και η φυστάμενη συνεργασία μας στο πλαίσιο της φυστάμενης εμπορικής, ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης έχει συμβάλει στην εξάλληψη ε, της φτώχειας στην ειρηνευτική διαδικασία και στην ενσωμάτωση των χωρών και στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, παρότι θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τις επιτυχίες μας, δεν θα πρέπει να απέχουμε από μία ειλικρινή αυτοκριτική ε, και να πούμε ότι η συμφωνία και η εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ δεν έχει επιφέρει όλα τα αποτελέσματα που επιθυμούσαμε. Οπότε ακριβώς αυτή η νέα εταιρική σχέση στη συνέχεια της νέας ε, συμφωνίας ε, Κοτονού αποτελεί μια ευκαιρία για την εκ νέων ίσχυση αυτής της ε, αυτών των προσπαθειών. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία θα είναι πιο ευέλικτη, πιο στοχευμένη και θα μας βοηθήσει να ε, βρούμε την άποψη προς τα μπροστά. Γι' αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την υφιστάμενη Γενική Συμφωνία με τρεις συμπληρωματικές περιφερειακές συμφωνίες για την Καραϊβική και, ε, και τον Ελληνικό η γενική συμφωνία ε, που καλύπτει δηλαδή όλες τις χώρες ε, θα πρέπει να είναι πιο ελαφριά. Αν θέλετε θα πρέπει να θέτει τους γενικούς στόχους, τις γενικές προτεραιότητες και να ορίζει κοινέ αξίες, συμφέροντα και τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας ε, στο παγκόσμιο πλαίσιο. Ε, βασιζόμενες τώρα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, οι τρεις περιφερειακές συμφωνίες θα πρέπει να ενισχύσουν, να ενισχυθούν και να επεκταθούν ουσιαστικά με νέες προτεραιότητες αλλά και με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ε, περιφέρειας. Επίσης συμφωνούμε μαζί σας ότι θα πρέπει να, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία ε, οι περιφερειακές, υποπεριφερειακές και τοπικές ε, οργανώσεις και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μία σειρά αποζητήματα για να στεφτούν με επιτυχία αυτές οι περιφερειακές συμφωνίες. Όπως και το Κοινοβουλίο θεωρούμε και εμείς ότι η εταιρική σχέση θα πρέπει να κατοχυρηθεί μέσω μιας δεσμευτικής ε, συμφωνίας. Γιατί ε, κάτι τέτοιο μας ε, διασφαλίζει περισσότερα πλέον εκτήματα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά δηλαδή συμβατικές υποχρεώσεις για, την, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργήσουμε σχέσεις ε, να εδραιώσουμε σχέσεις με περαιτέρω χώρες ε, με τις οποίες έχουμε κοινά συμφέροντα, ειδικότερα τις ε, χώρες της Βορείου αλλά και τις λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες και τις νησιωτικές χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην ομάδα κρατών ΑΚΕ. Με τη συμπερίληψη λοιπόν τέτοιων χωρών μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερο αντίκτυπο και περισσότερη συνοχή πολιτική σε ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Πέρα λοιπόν από τη συμπερίληψη νέων χωρών θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων των ε, ε, ενδιαφερόμενων των συναρμόδιων φορέων και δημοσίων και ε, μη δημοσίων σε περίπτωση εθνικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, φορείς του, του ιδιωτικού κλάδου. Και αυτή η εταιρική σχέση προφανώς θα πρέπει να λάβει και την κατάλληλη θεσμική υποστήριξη, έτσι ώστε οι αποφάσεις σε σχέση με τις ε, προγραμματισμένες δράσεις ε, να αναβάνονται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Τώρα χρειαζόμαστε μια συμφωνία η οποία θα έχει στον πυρήνα της το θεματολόγιο του 2030. Να έχουμε μια εταιρική σχέση η οποία πραγματικά ε, θα αφορά μια σχέση μεταξύ ομοτήμων. Και Επιτρέψτε μου να αναφερθώ συντομία στο τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξή. Όπω γνωρίζετε, η Συμφωνία Κοτονού θα εκπνεύσει το Φεβρουάριο του 2020, που σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν το 2019. Οπότε εγώ ε, θα διασφαλίσω ε, τη λήψη της κατάλληλης εντολής από το Συμβούλιο μέσα στο 2017 και με βάση την κοινή αντίληψη ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε ένα κοινό ε, κείμενο σε ό,τι αφορά δηλαδή μια δήλωση από την πλευρά μας μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2017. Μέσα στους επόμενους μήνες θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με το Συμβούλιο έτσι ώστε να υιοθετηθεί ε, το κείμενο αυτό της ε, νέας κοινή αντίληψης στο Συμβούλιο της 19ης ε, Μαΐου του 2017. Με αυτή την οριστική ε, την οριστικοποίηση ε, της ε, κοινή αντίληψης. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε τον Ιούνιο το κείμενο της νέας συμφωνίας και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε συγκεκριμένους στόχους για το επόμενο πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη. Και σε αυτή τη διαδικασία βέβαια το Κοινοβούλιο καλείται να παίξει όπως πάντα ένα ισχυρό ρόλο, δηλαδή να διασφαλίσει ότι ο ηγετικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι μόνο λόγια αλλά θα είναι πραγματικές πράξεις αναμένω με ενδιαφέρον την επικοδομητική συνεργασία από την πλευρά σας και τα σχόλιά σας και στο πλαίσιο βέβαια και της σημερινή συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Εμείς προσπαθούμε στα πλαίσια του χρονικού πλαισίου και οι συντονιστές ε, συμφώνησαν ότι το πρώτο εξάμεινο του 2017 θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν την διαδικασία εμείς ε, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας τώρα στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων και των στρατηγικών μας και όχι στον σχολιασμό τους ομόνων. Έτσι θα μας πάρουν σοβαρά τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάρουμε πρώτα τα σχόλια ή θα πρέπει να περιμένουμε και τις επόμενες δύο ανακοινώσεις να γίνουν εταιρική σχέση μετά το κοτονού, post κοτονού. Ίσως θα πρέπει να πάρουμε ε, με ξεχωριστό τρόπο απαντήσεις γιατί και οι δύο ανακοινώσεις έχουν μεγάλη σημασία. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Νόιζα. Βλέπω ότι είναι εδώ και η κυρία Κίνγκα. Ευχαριστώ πολύ Λίντα ε, και τον κύριο Επίτροπο για την παρουσίαση των ανακοινώσεων. Ε, βρισκόμαστε πάρα πολύ καλά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά μας ε, και ε, έχουμε το θέμα της απόφασης του Κοινοβουλίου αλλά και την ανακοίνωση όπου υπάρχουν ελάχιστες διαφορές τώρα. Στο προσκήνιο θα έλεγα ότι έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά ε, και ε, φαίνεται από το αποτέλεσμα ιδιαιτέρως αν λάβουμε υπόψη μας ότι αρκετά κράτη-μέλη ε, όσον αφορά την συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΑΚΕ ήταν διστακτικά. Έτσι λοιπόν και η Κομισιόν αλλά και το Κοινοβούλιο έπρεπε να ασκήσουν ε, ε, αρκετά, αρκετή δουλειά ώστε να τους πείσουν. Ε, επίσης, καταλαβαίνουμε ότι η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή και απέφερε πολλά διότι βασιζόμαστε σε αρχές οι οποίες δεν άλλαξαν ιδιαίτερως σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει δραματικά και νομίζω ότι σε αρκετούς τομείς ε, δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τόσο πολύ αυτές τις αρχές. Ιδιαίτερα όσον αφορά την κινητικότητα ε, των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, Επίσης όσον αφορά τη συνέχιση της συγκεκριμένης συμφωνίας θελήσαμε να συνδέεται άμεσα με την οικονομία αυτό και είναι σημαντικό το ότι και εσείς αλλά και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο αναγνωρίζουμε ε, την ε, σημασία της ε, Συμφωνίας Κοτονού και ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε περαιτέρω πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης είναι καλό το ότι εκπροσωπούμε και οι δύο τις άποψης ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική και τέλος θα ήθελα επίσης να προσθέσω όσον αφορά ε, την κατάσταση μετά την εκλογή του Τραμπ ε, βλέπουμε ότι στρέφεται η πολιτική προς ε, τον εαυτό της ε, και απομακρύνεται από, την, από το διεθνές. Είναι λοιπόν η σωστή κατεύθυνση αυτή που προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μέσω διεθνών συμφωνιών και να κάνουμε πρόοδους από κοινού ιδιαιτέρως προς συμφέρον των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών Επίσης καλό είναι ότι θα συμπεριλαμβάνεται και μια στρατηγική όπου θα συμπεριλαμβάνουμε τους ε, στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης για μέχρι το 2030. Ευχαριστώ λοιπόν ε, για την ανακοίνωση. Βρισκόμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος και θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο αποφασισμένα το επόμενο έτος για να πείσουμε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ωραία κάποιος άλλος ε, σχετικά με την συνεργασία μετά το Κοτονού, η κυρία Χόιμποκ. Ευχαριστώ ε, Λίντα, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Υπάρχουν πολλά στοιχεία σε αυτή την ανακοίνωση ε, που μπορούμε να υποστηρίξουμε, όμως υπάρχουν κάποια σημεία όπου έχω τις αμφιβολίες μου. Αναφέρεται για παράδειγμα ότι το ζήτημα της ε, μετανάστευσης ε, θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο όπως είναι για παράδειγμα η προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης, η δημοκρατία η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των κλιματικών αλλαγών. Όμως ανησυχώ λιγάκι διότι επιβαρύνουμε τον πολιτικό μας διάλογο με τους εταίρους μας με όλο αυτό το εύρος θεμάτων όπως είναι το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φιλών και ούτω καθεξής και γνωρίζουμε επίσης ότι ο διάλογος σχετικά με την μετανάστευση δεν ε, ε, βελτιώνει την κατάσταση σχετικά με τις παράνομες ροές προσφύγων και μεταναστών θα πρέπει λοιπόν ε, ε, να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη ε, συμφωνία σχετικά με την επιστροφή μεταναστών. Θα ήθελα μια ξεκάθαρη θέση για αυτό και ανησυχώ επίσης και για το σημείο όσον αφορά την ιδιωτική οικονομία και τη σύνδεση του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν αναρρύθμιτα παραδείγματα όπου πολυεθνικές δεν φροντίζουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες, ενδιαφέρονται μονάχα ε, για το δικό τους κέρδος, έχουν υπερεκμεταλλευτεί τους σπόρους, έχουν αφήσει πίσω τους ε, περιβαλλοντικές καταστροφές ε, άφησαν τους ανθρώπους σε άθλια κατάσταση επειδή δεν έχουμε το νομικό πλαίσιο για όλο αυτό και ε, επίσης και σε αυτή την ανακοίνωση δεν βλέπω να συμπεριλαμβάνεται το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και αυτό θα ήθελα να το σκεφτούμε και αυτό. Θετικό θεωρώ επίσης ότι συμπεριλαμβάνεται την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής τις προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως επίσης και ζητήματα που αφορούν ε, την φοροδιαφυγή, την απάτη. Όλα αυτά τα υπογραμμίζουμε και τα υποστηρίζουμε. Όσον αφορά τώρα την γεωργία, Εκεί θα μπορούσαμε ίσως να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά ε, την ε, γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν ε, διάφορα συστήματα. Χθε στην Επιτροπή Γεωργίας είχαμε έναν ειδικό ο οποίος δραστηριοποιείται ιδιαίτερο στην Αφρική και προσπαθεί να δημιουργήσει άλλα συστήματα όπως είναι ή να συνδυάσει τη γεωργία με την δασοπονία Προς αυτή την κατάευθυνση ε, πιστεύω ότι θα μπορούσαν ε, να συμπεριληφθούν όταν βλέπουμε την κατάσταση στην Αφρική. Λοιπόν, κατανοούμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα. Έκπληξη ε, είναι για μένα το ότι δεν περιλαμβάνουμε τίποτα ε, για τα γενετικά τροποποιημένα και έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς στο Κοινοβούλιο ότι δεν το υποστηρίζουμε αυτό, ιδιαίτερως βλέποντας τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις χώρες όπου έχουν εφαρμοστεί αυτά. Απογοητεύομαι επίσης διότι αναφερθήκατε στη συνεργασία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΑΚΕ σε πολυμερές επίπεδο, όμως αυτό το οποίο ε, θεωρώ ότι απουσιάζει είναι μια πρόταση σχετικά με το πώς μπορούμε να το προωθήσουμε όλο αυτό και να ε, υποστηρίξουμε τα κοινά μας συμφέροντα ε, σε αυτά τα πολιτικά επίπεδα. Και το βλέπω ως μια αντίφαση επίσης ως βασικό αίτιο αναφέρατε για ποιο λόγο δεν επιθυμούμε να έχουμε τρεις διαφορετικές συμφωνίες που να είναι δεσμευτικές ένας λόγος είναι ότι δεν έχουμε την, την ε, σκέψη να συνεργαστούμε σε ε, πολυμερή φόρα. Όμως ταυτόχρονα υπήρχε και η κριτική ότι όλο αυτό δεν έχει λειτουργήσει, διότι σε αυτά τα φόρα δεν ε, παρουσιαζόμαστε από κοινού με τις χώρες ΑΚΕ. και ο ίδιος μάλιστα συνειδητοποιήσατε ότι υπάρχει δυνατότητα για μια πιο ευέλικτη ε, διαθεσμική συνεργασία το ερώτημα λοιπόν που θέτω είναι πώς θα γίνει όλο αυτό, στην πρακτική πώς θα λειτουργήσει, διότι αυτό ακριβώς ήταν το σημείο το οποίο ως και τώρα δεν λειτουργούσε καθόλου. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλο αυτό το ε, πλαίσιο, όμως ε, θέλουμε να ενισχύσουμε αυτόν ακριβώς τον τομέα και να συνεργαστούμε περαιτέρω ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Ε, πιστεύω ότι χρειάζονται τρεις ισχυρές, ισχυρές συμφωνίες που θα βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα είναι δεσμευτικές και αυτή πιστεύω θα είναι η καλύτερη προσέγγιση. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και που κάθε τόσο έρχεστε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ και πριν δώσω το λόγο ε, στην ε, κυρία Κίνγκ θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Γενικό, τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης για, ο οποίος ήρθε να δεχθεί σχόλιο και να συμμετάσχει στη συζήτηση. Ε, κυρία Κέγγε, ευχαριστώ τον Επίτροπο να υπογραμμίσω κάποιες πλευρές από τις συμφωνίες μετά Κοτονού. Καταρχάς θα συμφωνήσω με το ότι το να υπάρχει μια νέα δεσμευτική συμφωνία είναι κάτι το θετικό. Ε, το επόμενο θέμα είναι η κοινοβουλευτική διάσταση. Εμείς έχουμε ανάγκη να διατηρήσουμε την κοινοβουλευτική αυτή διάσταση προσπαθώντας να την απομακρύνουμε από τον αυστηρά συμβουλευτικό χαρακτήρα της. Να υπάρξει μια γνωμοδότηση μένα, αλλά μια σημαντική γνωμοδότηση που θα επιτρέπει από τους διάφορους βουλευτές να αντιπαρατίθενται όπως πάντα το έκαναν με θετικό και επικοδομητικό τρόπο στα πλαίσια των συζητήσεών μας. Μια άλλη διάσταση τώρα, πολιτική διάσταση, την υπογράμμισαν οι συνάδελφοι σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, με τα θέματα των πολιτικών σχέσεων με τις χώρες ΑΚΕ. Το 8ο άρθρο σχετικά με τον πολιτικό διάλογο. Θα πρέπει να διατηρηθεί ο διάλογος αυτός και με τις υπόλοιπες χώρες. Κάτι τέτοιο θα μας επέτρεπε ίσως να προλαμβάνουμε κάποιες από τις συγκρούσεις, από την άλλη θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε την πορεία επικοινωνίας με τις χώρες αυτές, οι οποίες πολλές φορές παρουσιάζουν μια κάποια αστάθεια πολιτική. Τα άρθρα αυτά επιτρέπουν στα θεσμικά μας όργανα λοιπόν να εντάσσονται στο εσωτερικό ενός νομικού πλαισίου, που μας δίδει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις σχέσεις με τις χώρες αυτές. Αυτό το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Παράδειγμα είναι το Μπουρούντι, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, αφορμές. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν μιας επιπλέον μορφής προσοχής. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. θα υπάρξει ένα πλαίσιο και μέσα θα υπάρξει μια γεωγραφική κατανομή, περιφερειακή κατανομή. Ε, Καραϊβική, Ειρηνικός, Αφρική. Και για κάθε περιφέρεια εμείς θα ξεχωρίζουμε το ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. και για το εμπόριο. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε προβλήματα σε κάποιου τομεί τώρα. E Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα λοιπόν και με την Ανατολική Αφρική. Τώρα υπήρξαν κάποιε δυσκολίε με την Γκάνα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν έτσι και αλλιώς οι εμπορικές συμφωνίες γιατί το Κοτονού ασχολείται και με θέματα εμπορίου. Λοιπόν, μία απάντηση από τον Επίτροπο και μετά θα περάσω στον επόμενο εισηγητή. Ευχαριστώ τα αγαπητά μέλη για τις ε, ιδέες τους, τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους και τις ανησυχίες τους για το νέο πλαίσιο, το λεγόμενο μετά κοτονού. Να μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις τώρα ιδιαίτερα για την πορεία που θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Δεν θα τις χαρακτηρίσω καταληκτικές, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται και συμμετέχετε κι εσείς κι εμείς για να μπορέσουμε να ορίσουμε κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του 17 το διαπραγματευτικό μας πλαίσιο. Ξεκινώντας αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε ως Επιτροπή είναι να δούμε ποια είναι τα βασικά πλαίσια στα οποία θα σταθούμε για την επόμενη ε, ρύθμιση μετά κοτονού. Σχετικά με την ουσία της συγκεκριμένης πρότασης μπορεί κανείς να δει ότι πρόκειται για μια ουσιαστική μετακίνηση αυτό το οποίο προτείνουμε. Αντιθέτως από αυτά που ισχυρίζονται ορισμένοι εμείς δεν προτείνουμε την συνέχιση του ισχύοντος πλαισίου συμφωνίας Κοτονού, αλλά προτείνουμε πολύ σημαντικές αλλαγές. Ξεκινάμε καταρχάς από τα ειδικά χαρακτηριστικά ξεχωρίζοντας τις τρεις περιοχές ΑΚΕ, τις τρεις περιφέρειες ΑΚΕ και μετά πηγαίνουμε στο σύνολο των ΑΚΕ και όχι το αντίστροφο. Εμείς χρησιμοποιούμε την πραγματικότητα της ομάδας ΑΚΕ για να θέσουμε κανόνες και στόχους οι οποίοι να συμβαδίζουν με τα συμφέροντά μας τα συμφέροντά μας στα πλαίσια της Συμφωνίας του Κοτονού διευκρινίζονται σε, με σαφή τρόπο σε επίπεδο συμφωνίας στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου, της στήριξη των κανόνων του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής διακυβέρνησης, άρθρα 96, 13, 8, Είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτεί κανείς με 79 μεμονωμένες χώρες ε, τι δεσμευτικές, ε, αν θέλετε, πλευρές των ε, συζητήσεων. Γι' αυτό λοιπόν η πρότασή μας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να καταλήξουμε σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ή καλύτερα σε μια συμφωνία η οποία να βασίζεται σε κανόνες. Και η αντιμετώπιση αυτού του τύπου βρίσκεται ακριβώς, είναι ακριβώς ο πυρήνας της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολλές οι εμπορικές συμφωνίες τις οποίες έχουμε στον κόσμο και στα πλαίσια των οποίων εφαρμόζουμε τη συγκεκριμένη αυτή αντιμετώπιση. Το δεύτερο θέμα. Στα πλαίσια των συζητήσεων τις οποίες μέχρι τώρα είχαμε με την ομάδα ΑΚΕ και με τη Γραμματεία αλλά και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και τους σε επίπεδο υπουργών, συμβουλίου υπουργών κτλ. Καταλήξαμε στο ότι υπάρχουν ε, δύο ε, ισχυρές θέσεις, κεντρικές θέσεις για τη διαπραγμάτευσή μας για τη συμφωνία μετά Κοτονού. Η ομάδα αυτή καταρχάς τίνει στο να παραμείνει ενωμένη είτε εντός είτε εκτός της νέας συμφωνίας. Το δεύτερο κεντρικό σημείο είναι ότι η ομάδα ΑΚΕ θα προτιμούσε να έχει μια νομικά δεσμευτική σχέση με βάση συγκεκριμένους κανόνες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπ' αυτή τη λογική θα πρέπει όχι να προσπαθήσουμε σε όλα τα θεσμικά όργανα απλά να καταλήξουμε σύντομα σε μια διαπραγματευτική εντολή, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με τους εταίρους μας θέματα ουσίας και τις θέσεις, εν πάση περιπτώσει, τις οποίες έχουν για το τελικό πλαίσιο της συμφωνίας ή της ρύθμισης, αν θέλετε, μετά κοτονού. Έχει σημασία λοιπόν να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα σχόλια και κάποιες από τις απόψεις τις οποίες εκφράσατε μέχρι τώρα εδώ. Έχει σημασία ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα συνένεση, αλλά θα πρέπει και η νέα ρύθμιση να αντιμετωπίσει το θέμα της εταιρικής συμφωνίας του ιδιωτικού τομέα, της συμπερίληψης δηλαδή του ιδιωτικού τομέα στην εταιρική σχέση. Αν δούμε κανείς την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μέχρι τώρα, και αν δούμε το τι ισχύει σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές εταιρείες, μικρές, μεγάλες, ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι ε, από μόνοι τους, θα έλεγα, και επί τη βάση των δικών τους εμπορικών δραστηριοτήτων εμπλέκονται ε, στις χώρες ΑΚΕ. Μια εμπλοκή η οποία τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται και να έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Γενικά στο ε, χαμηλότερο επίπεδο, αν θέλετε, της προστιθέμενης αξίας των μορφών παραγωγής. Λοιπόν, βασικός μας στόχος είναι η εταιρική σχέση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να οδηγήσει σε μια πραγματικά αναπτυξιακή εταιρική σχέση και παρουσία με τον ιδιωτικό τομέα, του ιδιωτικού τομέα. Αλλά κάτω από κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα έχουν εκ των προτέρων ξεκαθαριστεί. Όπως οι πρόσφατες προτάσεις ε, για το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο Εμείς θα πρέπει να αναμίξουμε τη συμφωνία που έχουμε σε επίπεδο επιδοτήσεων με τις δανειοδοτικές δυνατότητες των πιστοτικών ιδρυμάτων και με τα προγράμματα εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αηφόρου Αναπτύξεως. Δηλαδή, περιμένουμε στην ουσία νέες επενδύσεις και στην Αφρική και στην Ευρωπαϊκή γειτονία με αυτόν τον τρόπο. Επενδύσεις όμως οι οποίες θα είναι συμβατές με τα κριτήρια ODA που θα συνεισφέρουν δηλαδή στους στόχους της χιλιετίας και που θα συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη, θα συνεισφέρουν στην εκβιομηχάνηση και την καταπολέμηση του αποκλεισμού των οικονομιών των χωρών εταίρων. Στις διαδικασίες δημιουργίας αξίας οικονομικής έτσι ώστε να μην εκμεταλλευόμεθα απλά τις οικονομίες και τους παραγωγικούς πόρους των οικονομιών αυτών αλλά να δώσουμε, να εμφυσίσουμε θέμενη αξία σε αυτές. Διόλου εύκολο. Πάντως αξίζει τον κόπο και είναι μάλλον απαραίτητο να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην αναπτυξιακή αυτή εταιρική σχέση. Δεν είναι κάτι το οποίο προβλέπεται μόνο στην συνένεσή μας και στο νέο πλαίσιο το μετακοτονού, αλλά είναι και τμήμα της Ατζέντα 2030 και των τρόπων χρηματοδότησης των αποφάσεων για την ανάπτυξη που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Τίθεται λοιπόν εδώ το θέμα του ρόλου του ιδιωτικού τομέα και υπάρχει επίσης και το ότι ένα από τα προβλήματα σε επίπεδο εφαρμογής, ακόμα και επικύρωσης της συμφωνίας αυτής, είναι ότι η συμφωνία συγκεντρώνει κυρίως την προσοχή της σε εμπορικές ρυθμίσεις, σε ρυθμίσεις πρόσβασης σε αγορές, και όχι στην προσπάθεια βελτίωσης της παραγωγικής αλυσίδας και αύξησης της προστιθέμενης αξίας των δυνατοτήτων των προϊόντων της παραγωγής των χωρών αυτών όπου θα ήταν κάτι τέτοιο πραγματική ε, ενίσχυση, βοήθεια. Στα πλαίσια λοιπόν της νέας συνένεσης και στα πλαίσια της νέας συμφωνίας μετά Κοτονού θα δοθούν οι δυνατότητες για μεγαλύτερη ανάπτυξη, για περισσότερη παραγωγή, για περισσότερη ε, ε, οικονομική δυνατότητα και βιομηχανική ικανότητα των χωρών αυτών, κάτι το οποίο θα επηρεάσει συνολικά τις εμπορικές μας απόλυτες με τους εταίρους μας στις χώρες ΑΚΕ. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο κονσένσου στην κοινή αντίληψη. Έχουμε δύο συνεισηγητές ε, εδώ, οι οποίοι πολύ πρόσφατα επέβαλαν την ε, έκθεσή τους ε, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, οπότε ε, καταρχήν ο λόγο στον κύριο και στη συνέχεια στον κύριο Νόζα. Ευχαριστώ ε, και χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι εδώ Επίτροπε και μάλιστα μία μόλις εβδομάδα μετά από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης από την πλευρά της Επιτροπής μαζί με τον ε, συνάδελφό μου, τον Νόρμπερτ Νόιζερ. Εμείς ε, συντάξαμε μία έκθεση στην οποία διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία που έχετε συμπεριλάβει στην ανακοίνωσή σας ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας απόψεις. Ε, με άλλα λόγια, ορίζουμε με τον ίδιο τρόπο τις κύριες κατευθύνσεις που θέλουμε να ακολουθήσουμε στο επίπεδο ε, της ε, περαιτέρω συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ. Μαζί με τον συνάδελφο Νόιζερ θεωρήσαμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πραγματικά θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της εταιρικής ε, σχέσης συνεργασίας, αυτή δηλαδή η 17 στόχοι και η ονομασία SDGs είναι απολύτως απαραίτητη για αυτή τη συνεργασία. Ε, ειδικότερα το σημείο 9, δηλαδή η πράσινη φιλοπεριβαλλοντική ε, εκβιομηχανισμός ή μηχανοποίηση θα πρέπει ε, να ετονιστεί περισσότερο και ενδεχομένω να συνδυαστεί και με το μεταναστευτικό ζήτημα. Η δική μας τώρα έκθεση τονίζει μεταξύ άλλων την ε, χρηστή διαχείριση, την ε, ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή του, ε, των πολιτών σε αυτή τη συνεργασία και θεωρούμε πως αποτελούν προτεραιότητα σε αυτές τις συμφωνίες αυτά τα ζητήματα όπως τα αναφέρετε κι εσείς αλλά δεν θα έπρεπε να τονιστούν ακόμα περισσότερο και να αναφέρονται ρητά δηλαδή αναφέρουμε ότι θα πρέπει να ε, υπάρξει ε, δέσμευση σε ό,τι αφορά τις ε, ενισχύσεις και θα πρέπει να αναπτυχθούν και οι κατάλληλες εταιρικέ σχέσει ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Στη δική σα ανακοίνωση γίνεται και, γίνονται και προτάσει σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτική μίσθωση, το leasing. Ναι, είναι σωστέ αυτέ οι ιδέε, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο εμφαντικοί, ώστε να υποστηρίξουμε περισσότερο την αμοιβαία συνεργασία τέτοιου είδους ε, αναφορές ε, δεν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει τέτοιου αναφορές να γίνονται συγκεκριμένα μέσα στην ανακοίνωση. Ε, σε ό,τι αφορά δικότερα τις εταιρικέ σχέσεις, νομίζω πως θα πρέπει να αναφερθείτε περισσότερο στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις των εργοδοτών ή την ακαδημαϊκή κοινότητα. θα πρέπει επίσης ε, να περιγραφεί ε, πιο συγκεκριμένα ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων, εάν πραγματικά προβλέπουμε ένα ρόλο για τα Εθνικά Κοινοβούλια, στο πλαίσιο δηλαδή της ε, διαμόρφωσης των εθνικών πολιτικών των σχετικών χάρων. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, ο Νόρμπερτ Νόιζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Μπόκταν. Πράγματι υπάρχει μια συνένεση μεταξύ μας σε ό,τι αφορά το consensus, την κοινή αντίληψη και μεταξύ μας ως ε, συζητητές, οπότε απλώς θα συμπληρώσω κάποια στοιχεία τα οποία κατά την άποψή μου είναι σημαντικά. Κατά δική μου λοιπόν άποψη θα πρέπει να τονίσουμε ε, περισσότερο ότι είναι αναγκαία η συνοχή των ε, πολιτικών και ενδεχομένω θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για αυτή την ανάγκη συνοχή τη πολιτική. Επίση ε, θα πρέπει να αναφέρουμε εμφατικότερα τι βασικέ μα αρχέ. Ναι, αναφέρονται ήδη, αλλά θα πρέπει ενδεχομένω να τονίσουμε περισσότερο την καλή συνεργασία, τον εκδημοκρατισμό, την εταιρική σχέση και το ρόλο τη κοινωνία των πολιτών. Αυτό ειδικότερα ε, σε σχέση με την ατζέντα του 2030 είναι σημαντικό. Δηλαδή να τονίσουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, γιατί χωρίς τη συμμετοχή της δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους σχετικούς στόχους. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να τονίσουμε και ε, τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Και αυτές αναφέρονται μεν, αλλά καλό θα ήταν να τονιστούν ακόμα περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ισχυρή ε, η μεγάλη έμφαση στη διαφάνεια και θα πρέπει να αναφερόμαστε ε, στα ωφέλη που αποκομίζουμε από ιδιωτικέ επενδύσεις όταν αυτά τα ωφέλη αφορούν πραγματικά τους ίδιους τους πολίτες, τους ε, πληθυσμούς αυτών των χώρων. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα το επενδυτικό σχέδιο, το Box Investment Plan, και πάλι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε τη διάσταση τη διαφάνεια και ειδικότερα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να αναλάβουμε μεγαλύτερο μέλο τη ευθύνη. Δηλαδή θέλουμε πραγματικά να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερε ελεγκτικέ διαδικασίε και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να αναλάβει ένα ρόλο παρατηρητή, observer, τόσο σε ό,τι αφορά τα καταπιστευματικά ταμεία και σε ό,τι αφορά το planning και ε, σε, αυτό το, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα ενδεχομένως θα, ε, να υπάρξουν κάποιες δαμάχες μεταξύ μας. Επίσης, ό,τι αφορά το Νταγκαμπελίτη, ενδεχομένως ε, ίσως θα πρέπει να διευκρινιστεί λίγο το τι ακριβώς εννοούμε με τις ε, στρατιωτικές δράσεις, military actions. Ίσως θα πρέπει να έχουμε και πιο σαφείς ορισμούς δηλαδή σε σχέση με αυτές τις έννοιες, γιατί εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσουμε την το ελεγκτικό μας δικαίωμα, ε, την εξουσία που έχουμε. Νέος στόχος του 0,7% του ε, εθνικού εισοδήματος είναι ε, σωστός, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το κράτη θα ανταποκριθούν σε, αυτόν τον, σε αυτή τη δέσμευση. Και από εκεί και μετά να πω ότι χθε εδώ είχαμε προσκεκλημένο τον ειδικό ε, απεσταμμένο των Ηνωμένων Εθνών, τον David Ναμπάρο, για τα ζητήματα βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, των ΗΠΑ, ο οποίο ε, συνεχάρει την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για τη δουλειά που κάνουν σε αυτό το τομέα. Οπότε θεωρώ πω ε, βρισκόμαστε στο κατάλληλο χρονικό σημείο. Είναι σωστή χρονική συγκυρία για τη δημοσίευση αυτών των δύο ανακοινώσεων τη Επιτροπή. Και να πω και κάτι άλλο που είπε ο κ. Ναμπάρο χθε. Εάν, εάν δεν θέλουμε να υπάρχει πλέον διαχωρισμός μεταξύ των ανεπτυγμένων εντό εισαγωγικών χωρών και των αναπτυσσόμενων χωρών, αν δηλαδή είμαστε όλε υπό ανάπτυξη χώρε ε, σε σχέση ακριβώ και με την ατζέντα του 2030, τότε ε, θα πρέπει να, έχουμε, να αναλάβουμε και ως επιτροπή, κοινοβουλευτική επιτροπή, μια άλλη ονομασία. Ε, δηλαδή, θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με εμάς τους ίδιους και να σκεφτούμε πώ μπορούμε με την αλλαγή, για παράδειγμα, τη ονομασία τη επιτροπή μα να δώσουμε το έναυσμα προ αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την ίση μεταχείριση σε αυτό το επίπεδο, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ανάπτυξη των διαφορετικών χώρων. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο η Μαρία Χόιμπουχ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ένα ε, μόνο ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Ε, η κοινή αντίληψη έχει ένα πολύ μεγάλο χρονικό ορίζοντα, έως το 2030 δηλαδή. Και πέρα από την προτεραιότητα της καταπολέμησης της φτώχειας, η οποία ευτυχώς βέβαια έχει παραμείνει μέσα ε, σε αυτή την κοινή αντίληψη και στην οποία θα δοθεί και προτεραιότητα, αναφέρονται ε, και η ασφάλεια και η καταπολέμηση της η πρόληψη της μετανάστευσης. Ε, άρα λοιπόν με βάση αυτό το μεγάλο χρονικό ορίζοντα σκέφτομαι πώς θα γίνει αυτή η κατανομή, αν θέλετε, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων θα παραμένει πραγματικά κύρια προτεραιότητα η, καταπολέμηση της φτώχειας ή θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην ασφάλεια και το μεταναστευτικό ζήτημα. Ε, πρόεδρος. Νομίζω πως ε, σε ό,τι αφορά τον κύριο στόχο του εγγράφου θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ε, θέλουμε να υπάρχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ της, ε, του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή, γιατί είμαστε ο μεγαλύτερο χορηγό ε, παγκοσμίω. Οπότε θα πρέπει να, έχουμε, να διασφαλίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο αυτή τη ε, βοήθεια και τη ενίσχυση που παρέχουμε. Ένα όμω ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι το εξή. Τι είναι αυτά τα box, γιατί σε τι χρησιμεύουν. Δηλαδή είναι αρκετά μακροσκελέ το κείμενο, αλλά υπάρχουν αυτά τα boxes εδώ, αυτά πλαίσια, αν θέλετε, κάποια κουτάλια δηλαδή μέσα στο κείμενο. Συνήθως αυτά περιλαμβάνονται για να εξηγήσουν ε, κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο ή κάποια πτυχή του κονσένσου. Οπότε ένα ερώτημα έτσι, απλά από την πλευρά μου. Σε τι χρησιμεύουν αυτά τα πλαίσια. Γιατί βέβαια οι διαπραγματεύσει μας αποτελούν ε, ε, αφορούν αυτό το έγγραφο. Οπότε το τι περιλαμβάνει σε αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό. Και με τι ακριβώς είναι αυτά τα πλαίσια, τι περιλαμβάνει σε αυτά. Ευχαριστώ για ε, τις απόψεις, τις συνεισφορές σας στην όλη συζήτηση όσον αφορά τη συνένεση για την ανάπτυξη ε, αυτή θα καθορίσει τις ε, δράσεις ε, ανάπτυξης ε, και θα συντονίσει καλύτερα το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών εν ώψη των, της Ατζέντα 2030 για τους αναπτυξιακούς στόχους, τους βιώσιμους στόχους. Τόσο, τώρα όσον αφορά το κείμενο της συνένεσης, είναι, έχει μια ενιαία εικόνα και είναι ένα ε, κείμενο το οποίο αναφέρεται σε όλα τα ε, σχετικά και σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν αναφερθεί και σήμερα εδώ από εσάς. Υπάρχουν όλα μέσα στο κείμενο, όμως ε, συνεχίζουμε τη συζήτηση ούτως ώστε να έχουμε μια ε, κοινή συνένεση εξετάζοντας τώρα ε, την ίδια τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο ε, κείμενο ορισμένες από τις ε, οδηγίες και κατευθυντήριες θα μπορούσαν να, να είναι με έναν πιο ξεκάθαρο τρόπο γραμμένες Επίσης πρέπει να ε, παρατηρήσουμε ότι όσον αφορά το συνολικό κείμενο της ε, συνέντησης υπάρχει μια ξεκάθαρη ε, υπάρχουν ξεκάθαρες προτεραιότητες μέσα σε αυτό όσον αφορά τις αναπτυξιακές μας δράσεις. Μεταξύ αυτών είναι η καταπολέμηση της φτώχειας που βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Υπάρχει ένα ευρύτερο λοιπόν πλαίσιο για την καταπολέμηση της φτώχειας ε, και για τον βιώσιμο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να ε, αντιμετωπίσουμε τα αναπτυξιακά ζητήματα στην παγκόσμια ατζέντα. Και γι' αυτό τον λόγο προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία κατά πολέμηση της φτώχειας, ε, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα όλες, ε, όλα τα εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης για να μπορέσουμε να ε, επιτύχουμε το συγκεκριμένο στόχο. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε και το γενικότερο πλαίσιο διότι υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας πάνω στον οποίο ε, συνδέονται όλα αυτά, δηλαδή ε, η ανάπτυξη και η μετανάστευση, η ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια, ε, η ανάπτυξη και η ασφάλεια. Το πλαίσιο λοιπόν της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι πολύ πιο ευρύ σε σχέση με την παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια που ορίζεται από τις δυνατότητες των αναπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε ε, την, ε, το σημείο συνάντησης όπου θα φέρουμε τις δικές μας δράσεις ανάπτυξης για να μπορέσουμε ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τους λοιπούς αναπτυξιακούς στόχους οι οποίοι σχετίζονται με τη μετανάστευση για παράδειγμα ή την ε, ασφάλεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προσέγγιση που προτείναμε ε, στο consensus ε, λαμβάνει υπόψη όλες τις δράσεις και στον τομέα της μετανάστευσης αλλά και σε αυτόν της ασφάλειας όπου χρησιμοποιούμε εργαλεία σχετικά με την ανάπτυξη τα οποία ταιριάζουν με τις δράσεις του ODA. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ταυτόχρονα ότι τα ε, κριτήρια αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο ευρύτερο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Υπάρχει λοιπόν μια ατζέντα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και νέα κριτήρια ODA πάνω στα οποία θα πρέπει ε, να συμφωνήσουμε στον ΟΑΣΑ αλλά και στην Επιτροπή ΝΤΑΚ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στο σύνολό της μέλος εκεί, όμως τα περισσότερα κράτη-μέλη συμμετέχουν και θα πρέπει ταυτόχρονα να συντονίσουμε καλύτερα τις δράσεις μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε και να συμφωνήσουμε στον ΟΑΣΑ σχετικά με τα κριτήρια ODA τα οποία θα ε, συμπεριληφθούν σε όλο αυτό το ευρύτερο πλαίσιο ε, της ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη. Όσον αφορά τη σχέση ανάπτυξης και ασφάλειας, αυτή τη στιγμή δεν χρηματοδοτούμε με τα εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο στρατιωτικό εξοπλισμό ή εκπαίδευση ε, σε ιδιάζουσες περιπτώσεις ε, όπου υπάρχουν θεσμοί στις χώρες εταίρους ε, οι οποίοι δεν παρέχουν τα αναγκαία μέτρα, τότε εμεί ε, παρέχουμε μια κάποια εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού για να μπορέσουν αυτοί στη συνέχεια να συνεισφέρουν σε ζητήματα ασφάλειας, ε, υπό, τον, υπό το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτω ώστε ο στρατός να συνεισφέρει στην εσωτερική ασφάλεια αλλά και για να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για την ε, επιτυχημένη ανάπτυξη ε, σε, στην περίπτωση τέτοιων προγραμμάτων. Υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή λοιπόν αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ανάπτυξη και την ασφάλεια και ε, δεν περιλαμβάνει τον στρατιωτικό εξοπλισμό όταν το ζήτημα αφορά ε, την ε, χρηματοδότηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με την αναπτυξιακή συνεργασία. Επίσης, θέλουμε να δράσουμε με αναπτυξιακά μέσα και να ε, κινηθούμε με βάση τις ε, δύο βασικές ε, γραμμές που αφορούν το μεταναστευτικό πλαίσιο. Πρώτον, να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της μετανάστευσης και δεύτερον, να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση, το τράφικινγκ και να γίνει αυτή η μετάβαση από την παράνομη στην νόμιμη μετανάστευση και το κάνουμε ε, με ένα πλαίσιο το οποίο είναι σύμφωνο με το ODA. και το έχουμε επιβεβαιώσει και με βάση τα κριτήρια DAC του άσα Γενικότερα όμως είμαστε σε μια καλή φάση ε, και με το Συμβούλιο και με το ε, Κοινοβούλιο και με την ε, Κομισιόν ούτω ώστε να έχουμε μια κοινή ανακοίνωση και να υποστηρίξουμε μια τέτοια συνέντευξη μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς και πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όπως είναι για παράδειγμα η κοινωνία ε, των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας ε, και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς που μετάσχουν στην αναπτυξιακή συνεργασία όπως είναι η, αναπτυξιακή, η Τράπεζα Επενδύσεων και θα πρέπει να υιοθετήσουμε και να προσαρμόσουμε αντίστοιχα ε, το ευρωπαϊκό consensus το οποίο θα έχει την υποστήριξη και θα υπογραφεί από τη στιγμή που θα ε, λάβει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, ε, του Συμβουλίου και της Κομισιόν αλλά να έχει και την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα, ε, της κοινωνίας των πολιτών, άλλους, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, άλλους ε, ε, θεσμούς για να είναι ιδιαίτερα ισχυρό ώστε να ε, μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όταν το ζήτημα αφορά την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω όμως ότι ε, μας ξεφύγατε διότι ε, ο Άλλη με χαιρετάει από εδώ και θέλει να δηλώσει κάτι ακόμα. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερως για την κατάσταση σε σχέση με το ODA. Συζητήσαμε το θέμα με το Σουηδό Υπουργό και είπατε ότι υπάρχει μια επανατοποθέτηση του πλαισίου. Πότε θα ολοκληρωθεί η αναδιαρρύθμιση αυτή και ποια θα είναι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σαν παράδειγμα το κόστος της λήψης υπόψης, υπόψη της κατάστασης της μεταναστευτικής στις διάφορες χώρες είναι κάτι το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο γι' αυτό έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε αυτή την επανατοποθέτηση. Και ένα τελευταίο σημείο. Είπατε ότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. um, kind of uh, special... Σε σχέση με την ICSP Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σε σχέση με τους τρόπους χρηματοδότησης. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα γίνει. Κοιτάξτε, ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις και σε κάποιες από τις προηγούμενες. Καταρχάς, για τα λεγόμενα box. Ακριβώς αυτά τα θέματα είναι αυτά τα οποία διευκρινίζουν και συγκεντρώνουν την προσοχή μας σε συγκεκριμένα θέματα όπως εκπαίδευση, χώρες μεσαίου εισοδήματος, είναι οι λεγόμενοι δίκτες οι οποίοι ορίζουν το πεδίο με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε είναι πλήρως, ε, πλήρες τμήμα του κειμένου και βρίσκονται εκεί ακριβώς για να ε, υπογραμμίσουν τα θέματα τα οποία χρήσουν προσοχή. Για το ODA, γιατί έχω κληθεί επανειλημμένα να το σχολιάσω το θέμα αυτό. Συνεχίζεται η επανατοποθέτηση αυτή σε σχέση με το αντίστοιχο τάκ για τις ιδιωτικές επενδύσεις για το θέμα επίσης της μετανάστευσης, αλλά δεν έχει σε σχέση ε, με την επιλεξιμότητα των κονδυλίων για τα ΤΑΠ. Αυτά ήδη υπάρχουν. Δεν ξέρουμε τι μορφή θα πάρει αυτό, αλλά η θέση μας είναι δεδομένη και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη συγκεκριμένες δαπάνες ε, οι οποίες γίνονται σε ορισμένες χώρες για να δοθεί ενίσχυση στους μετανάστες. Τώρα, αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτούς που επιστρέφουν στις χώρες τους και την ενίσχυσή τους. Εδώ δεν έχουμε κάποιο κωδικό, δεν προβλέπεται ξεχωριστή κατηγορία. Και κάθε χώρα μέλος το θέμα αυτό το βάζει σε διαφορετικά κεφάλαια, θέσεις απασχόλησης, επανένταξη στην αγορά εργασίας κτλ. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν το εξής θέμα. Αν είναι δυνατόν τα κονδύλια τα οποία δίδονται στις χώρες προέλευσης για να βοηθηθούν οι πρόσφυγες ε, για να ενισχυθούν αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν στις χώρες τους θα πρέπει να δούμε αν ε, ε, όλα αυτά γίνονται με ικανοποιητικό τρόπο. Μιλάμε για δαπάνες οι οποίες γίνονται σε χώρες όπως η Σενεγάλη, το Μαλί κτλ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κωδικός DAC σε σχέση με αυτό και υπάρχουν κάποιοι επιπλέον κωδικοί οι οποίοι κάθε φορά δίδονται σχετικά αυθαίρετα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να καταστούν συμβατά με το γενικότερο ODA και τους κωδικούς. Γιατί όπως είπα εμείς προσπαθούμε να δαπανίσουμε κάποια κονδύλια στις χώρες προέλευσης έτσι ώστε να επαναντάξουμε τους ανθρώπους αυτούς να βρουν θέσεις απασχόλησης αλλά δεν υπάρχει μια γενικότερη ε, σύνδεση με κοινωνικού τύπου παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε εμείς στα πλαίσια ας πούμε της ε, ανταμετώπισης της ανεργίας. Αυτά για τη μετανάστευση, για το ICSP, από πού έρχονται τα 100 εκατομμύρια. Αυτό το συζητάμε ακόμα αλλά υποτίθεται ότι προέρχονται από επιπλέον πόρους, είτε από το ENI, είτε το PCI, που ανήκουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως και το IDF. Δεν έχουμε καταλήξει σε μια τελική συμφωνία. Πάντως η πρόταση είναι αυτή. Καλό συνάδελφε, θέλω να τελειώσουμε τώρα. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε άλλο, γιατί στις 11 έχουμε μια κοινή συνάντηση με την ΑΦΕΤ για την ανθρωπιστική κρίση στη Συρία και έχουμε δύο επιπλέον θέματα. Και από ό,τι φαίνεται εδώ ότι το <coughs> Αλεπί έχει ήδη πέσει στα χέρια της Συριακής κυβέρνησης. Το θέμα λοιπόν έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντική σημάντηση Έχουμε πολλούς ε, προσκεκλημένους, έχουμε και τον εκπρόσωπο της Ένωσης και 11 η ώρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τελειώσουμε εγκαίρως. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μίμητσα που ήρθε μαζί μας σήμερα. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτική η ε, προσπάθεια την οποία κάνουμε. Ευχαριστώ και τον Γενικό Διευθυντή. And of course at 3 o'clock we have our report back from the Council. Ε, και στις 3 ε, βέβαια θα έχουμε και την έκθεση από το Συμβούλιο και κλεισμένο των θυρών. Ε, συνάδελφοι, προσθέσαμε δύο ε, σημεία στην εμείς διάταξή μας ε, τα οποία είναι μεν σημαντικά, αλλά είναι σύντομα και αυτό γιατί όπως σας είπα θέλω να ε, διασφαλίσω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει ε, τα πάντα έως τις 11. Η επόμενη συνεδρίαση δηλαδή μαζί με την Επιτροπή ΑΦΕΤ, ε, σας πενθυμίζω, αιθουσα συνέδρια 2Q2. Okay, if those Αν αποχωρείτε, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε σιωπηλά γιατί έχουμε μία σειρά από σημεία ακόμα έως τις 11. Οπότε, σας παρακαλώ εδώ, ε, όσοι βρίσκεστε εδώ πίσω-πίσω στις σειρές, εδώ σας παρακαλώ, μην ε, κάνετε εδώ πηγαδάκια εντό εισαγωγικών. Αποχωρήστε από την αίθουσα αν θέλετε να μιλήσετε, γιατί πρέπει να αναφερθούμε καταρχήν στο θέμα του προπολογισμού. Πραγματικά πρέπει να προχωρήσουμε. Οπότε, περνάμε στο σημείο 9α, δηλαδή συμφωνία σε σχέση με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2017 έλαβε χώρα ο τριμερής διάλογος και η Επιτροπή προπολογισμού υιοθέτησε το αποτέλεσμα και ψήφισε επί αυτού του ε, φακέλου και αύριο, α όχι την πέμπτη, την πέμπτη στην Ολομέλεια λοιπόν θα γίνει η ψηφοφορία αυτού, του, αυτής της ε, συμφωνίας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ε, τι συμβαίνει, δηλαδή τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν ε, δηλαδή οι προτάσεις που είχαμε κάνει για τον προϋπολογισμό έγιναν δεκτές ή όχι, ο συγκεκριτής μου αυτό το ζήτημα είναι ο Νίτσι Ντέπα, οπότε θα του δώσω το λόγο και μετά στους υπόλοιπους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Πάντοτε βέβαια είναι, επιχαίρουμε το γεγονός ε, του να μπορούμε να, δώσουμε, ε, να επιστρέψουμε εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, και να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα του προπολογισμού είναι θετικά. Ε, όπως ήδη αναφέρθηκε στις 17 Νοεμβρίου οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου έφτασαν σε μια συμφωνία με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το τμήμα του προπολογισμού που αφορά τη δική μας εντολή, ε, υιοθετήθηκε ε, το σχέδιο της συμφωνίας ε, που είχε υποβάλει η Επιτροπή, αυξάνοντας όμως ε, σημαντικά δύο γραμμές του προπολογισμού σε συνέχεια και μιας επιστολής διορθωτικής από της Επιτροπής ότι αυτό το σχέδιο του προπολογισμού και αποτελεί πραγματικά, μας δημιούργησε κάποια έμπληξη στο ότι ξαφνικά μετά από την υποβολή του πρώτου σχεδίου τον Ιούλιο ήρθε τον Οκτώβριο η Επιτροπή για να ε, μας ζητήσει περισσότερη χρηματοδότηση και αντιλαμβανόμενοι πλέον το τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο ερχόμενοι σε επαφή με την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, ε, εδώ ενδιαφέρει το να δούμε το τι ζητήσαμε και το τι λάβαμε, λεπτομέρως. Με τις ε, τροποποιήσεις που έγιναν και το 21η Αυγούστου, ε, θέλουμε να ε, αναστραφεί αυτή η αυγουστου θελουμε να αναστραφει αυτη η ε, περικοπή του τάξη των 70 εκατομμυρίων ευρώ που είχε προτείνει το Συμβούλιο ε, σε ό,τι αφορά την αστροπηδική βοήθεια και να διατηρηθεί ε, και η υπόλοιπη χρηματοδότηση στα ίδια επίπεδα. Οι πιέσεις που είχαν ασκεθεί στις γραμμές του υπολογισμού σε ό,τι αφορά την αστροπιστική βοήθεια έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά από την προσφυγική κρίση και τα όσα συμβαίνουν στην ε, Τουρκία, στη Συρία ε, και αυτούς τους μεγάλους αριθμούς ανθρώπων που ζητούν ε, βοήθεια από εμά, αλλά και τους ανθρώπους που έρχονται από την Αφρική και διασύζουν τη Μεσόγειο. Η περικοπή λοιπόν που από το Συμβούλιο ήταν πραγματικά κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Ε, ένα λοιπόν δισεκατομμύριο 211 εκατομμύρια ζητήθηκαν. Δηλαδή γύρω στα 18 εκατομμύρια υψηλότερα από ό,τι είχε ζητήσει το Συμβούλιο για το 2017 αλλά σε συγκρίσιμα επίπεδα ε, με το, της περίοδου 2011-2016. Ε, και θέλαμε να αυξήσουμε το έκτακτο αποθεματικό κατά 20 εκατομμύρια. Ε, οι υπόλοιπε ε, ε, κατευθύνσει γραμμέ θέλουμε να μείνουν όπω προβλέπονται στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, όπω βέβαια είχε προβλέψει και η Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις γραμμές του προπολογισμού για την Ασία και τη Μέση Ανατολή, όπως και την ασφάλεια των τροφίμων. Εμείς είχαμε από τη δική μας ε, ζητήσει αυξήσει ανάλογε με αυτέ ε, του σχεδίου προπολογισμού στο σύνολό του και επίση θέλαμε να καταργηθούν οι περικοπέ ε, που είχε προβλέψει το Συμβούλιο για τη Λατινική και Νότια Αμερική και την ενίσχυση των οργανώσεων τη Κοινωνία των πολιτών. Ε, αντιδρώντας στην μεταναστευτική κρίση θέλαμε η να αυξηθεί η σχετική γραμμή του προϋπολογισμού κατά 7,1% ή 12,8 εκατομμύρια ε, ευρώ. Ε, εμείς είχαμε υποστηρίξει και ουσιαστικές ε, αυξήσεις της γραμμής του προϋπολογισμού της ανθρωπικής βοήθειας και η συμφωνία που επιτεύχθηκε προβαίνει σε μια αύξηση, η οποία βέβαια ε, δεν φτάνει τα επίπεδα που είχαμε ζητήσει, αλλά ξεπερνά σε κάθε περίπτωση το έκτακτο αποθεματικό. Επίση, η Επιτροπή Προπολογισμού υποστήριξε τι προτάσει που κάναμε σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, ε, τη γραμμή για το άσυλο και θέλησε να αυξήσει και την γραμμή για την Ασία ε, κατά 10 όμως εκατομμύρια ε, την αύξηση αντί για 44 εκατομμύρια όπως είχαμε προτείνει εμείς. Μετά λοιπόν δύο εβδομάδες μετά από την ε, ψήφο στην Επιτροπή Προπολογισμού και όπως σας είπα κάτι το οποίο μας δημιούργησε έκπληξη η Επιτροπή υπέβαλε ένα διορθωτικό του προπολογισμού γιατί προέβησε αύξηση δύο γραμμών του προπολογισμού για την Ασία και για τη μετανάστευση. Η γραμμή λοιπόν για την Ασία προτάθηκε προτάθηκε να αυξηθεί από 671 εκατομμύρια σε 771 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 100 εκατομμύρια ευρώ. Και ένα άλλο, ε, μια άλλη αυξήση που μα δημιούργησε έκπληξη, η γραμμή μετανάστευση. και η γραμμή λοιπόν για τη μετανάστευση να αυξηθεί από 48,2 εκατομμύρια ευρώ σε 448 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της άξης του 850%. Δηλαδή αυτό ε, καταδεικνύει ότι ξαφνικά ξύπνησε η Επιτροπή, ήρθε σε επαφή με την πραγματικότητα και είδε ποια είναι η απαραίτητη χρηματοδότηση για να αποκριθεί στους ε, στόχους των σχετικών γραμμών του προπολογισμού. Εμεί είχαμε ζητήσει αυξήσει και στι δύο γραμμέ του προπολογισμού, ε, πιο ισορροπημένο τρόπο. Αλλά ω Επιτροπή αρμόδια για αυτά τα ζητήματα από την πλευρά του Κοινοβουλίου, ίσω θα πρέπει να αναρωτηθούμε το τι συνέβη ανάμεσα στον Ιούνιο που ε, έβαλε η Επιτροπή το πρώτο σχέδιό τη έω τον Οκτώβριο για να αλλάξει με τόσο δραματικό τρόπο την άποψή τη και να προβεί ε, σε ε, μια τέτοια δραματική πρόταση. ιδιαίτερα αφού ε, ζητήσαμε από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα ζητήματα αυτά μετά από την υποβολή του πρώτου σχεδίου, αλλά ε, και στην ε, διαδικασία διαβούλευση. Οπότε πραγματικά είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι η Επιτροπή φάνηκε διατεθειμένη να επανεξετάσει τη θέση τη και να την αναθεωρήσει. Είχαμε ζητήσει περισσότερα κονδύλια σε ό,τι αφορά το DCI, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε σε ποιο, πώς θα αξιοποιηθούν τα κονθήλια τα οποία θα αξιοποιηθούν από το έκτακτο περιθώριο, το contingency margin. Και θα πρέπει να δούμε πώς ε, ακριβώς θα καλυφθούν τα compacts για τη μετανάστευση. Γιατί ένα πράγμα είναι το να λέμε ότι αυξάνουμε κατά δραματικό τρόπο την σχετική χρηματοδότηση, τα κονδύλια χρηματοδότησης και άλλο πράγμα είναι ε, το να ανταποκριθούμε στις, στα καθήκοντά μας σε σχέση αυτούς τους τομείς και πώς μπορούμε εμείς να ελέγξουμε ε, το πώς δαπανώνται τα σχετικά κονδύλια. Ναι, προφανώς είναι λίγο πρόωρο το να συζητήσουμε το πώς θα παρακολουθήσουμε αυτή την αξιοποίηση των κονδυλίων, αλλά νομίζω πως σε κάποια φάση θα πρέπει να συμφωνήσουμε έναν τρόπο ε, λειτουργίας, δηλαδή το τι ακριβώς θα κάνουμε για τον έλεγχο ως Επιτροπή Ανάπτυξης ε, και Επιτροπή ε, Προπολογισμού. Επιτύχαμε λοιπόν αυτές τις σχετικές ε, αυξήσεις στις δύο γραμμές του προπολογισμού. και συνολική αύξηση 834% για τις δύο γραμμές, δηλαδή τη μεταναστευτική και την ανθρωπιστική. Και είχαμε ζητήσει και περαιτέρω αυξήσεις σε σχέση με αυτές τις γραμμές και θα θέλαμε να ακούσουμε και από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ το πώς θα ανταποκριθεί με αυτά τα αυξημένα κονδύλια στις αυξημένες ανθρωπιστικές ε, προκλήσεις μέσα στα επόμενα χρόνια. Ε, το έκτακτο προθεματικό που παραμένει στα 315 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αυξημένο μόνο κατά, 4, ε, με κατά 6 εκατομμύρια, Ε, ακόμα και αν ε, αξιοποιηθεί στο σύνολό του αυτό το έκτακτο αποθεματικό θα υπάρξει μείωση της συνολικής ε, ε, χρηματοδότησης. Οπότε, από τη μία πλευρά επιχαίρουμε το γεγονός ότι στο πλαίσιο των μεταναστευτικών compact θα υπάρξει αύξηση της σχετικής γραμμής του προπολογισμού, αλλά στο σύνολο η χρηματοδότηση της υποστήριξη μέσω χρηματοδότησης ανθρωπιστικής βοήθειας θα είναι δύσκολη μέσα στο 2017. Ε, τέλος, θα θέλαμε να ζητήσουμε η Επιτροπή του Υποπολογισμού μέσω ενό διορθωτικού αυξημένε ε, πιστώσει ανάληψης υποχρεώσεων ε, στις ε, σχετικέ γραμμές μόλις θα εγκριθεί το αρχικό σχέδιο του προβλήσμου. Θα σταματήσω εδώ για να ακούσουμε και από την Επιτροπή το πώς ακριβώς ε, σκοπεύει να δαπανίσει αυτά τα χρηματοδοτικά κονδυλία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ναι, 8 ε, ε, λεπτά έχουμε μόνο στη διάθεσή μας ακόμα, γιατί μετά πρέπει να περάσουμε στο σύστημα για την Κολομβία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στο ζήτημα της Ασίας και της ε, μετανάστευσης, όμως όσον αφορά ε, τον έλεγχο της ροής των μεταναστών θα πρέπει να κάνουμε κάτι κατά τόπους ούτως ώστε να μην υπάρχει λόγος μετανάστευσης. Το ζήτημα της βοήθειας λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί. Έχουμε μία πρόταση λοιπόν ε, που είναι χαμηλότερη από το επίπεδο έναρξης ε, της πρότασης του 2016 για τον προϋπολογισμό και θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς μπορούμε να ε, προχωρήσουμε από αυτό το σημείο και καθώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε πάνω σε αυτό θα ήθελα να επαναλάβω και πάλι το ζήτημα των Trust Fund, Ταμείο Υπεραναπτυσσόμενων Χωρών. Θα έχουμε ε, μια ε, πρόταση ε, που θα περιλαμβάνει και αποστολές του Κοινοβουλίου, όμως μακροπρόθεσμα δεν θεωρούμε αυτό το εργαλείο καλό, διότι το Trust Fund για την Αφρική θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην δουλειά μας όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία έχει επιφέρει και δεν θα πρέπει να αφιερώνουμε τόσο πολύ χρόνο εξετάζοντας όλο αυτό, όμως ε, το έργο στο σύνολό του ε, ε, δεν συμφωνεί με το Κοινοβούλιο όπως το βλέπω εγώ. Η παρούσα είναι και η ε, Κομισιόν. Αρχικά έχουμε τη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω προσωπικά, να ευχαριστήσω επίσης και την Επιτροπή σας για την μόνιμη στήριξη την οποία μας παρέχετε στα πλαίσια μιας διαδικασίας δημοσιονομικής μακράς, δύσκολης, αλλά είναι σαφές ότι για την διεύθυνσή μας έχετε προσφέρει πολλά. Ε, χάρη στη συνεχιζόμενη λοιπόν προσπάθειά σας ε, όλα τα στοιχεία τα οποία δίδεται είναι συμβατά με τις προτάσεις που είχαμε καταρχάς κάνει. Είναι μεγάλη σημασία σε αυτό για να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική και να διαθέτουμε τα απαιτούμενα κονδύλια. Όπως υπόθηκε άλλωστε ήδη, καταθέσαμε μία πρόταση διορθωτική για τον προϋπολογισμό των υπαριθμών 1 και ζητήσαμε 150 εκατομμύρια από αυτά τα 150 εκατομμύρια μόνο 79 έγιναν δεκτά και το DCI αυξήθηκε επίσης κατά 457 εκατομμύρια. Όπως είπατε λοιπόν, η γραμμή μετανάστευσης η 357, με 357 και το άσυλο με 200 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει λοιπόν πώς διατίθεται τα χρήματα αυτά σε σχέση με τη μετανάστευση από την Βόρειο Αφρική και την Μέση Ανατολή. Πρόκειται λοιπόν για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Στα πλαίσια τώρα αυτής της διορθωτικής επιστολής του προϋπολογισμού έχουμε προτείνει 257 εκατομμύρια για το Ταμείο Εγγυήσεων και το Ταμείο Αηφορίας. Το Ταμείο αυτό δεν έχει ακόμα νομική βάση βέβαια, οπότε τα χρήματα δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα εκταπιεύσουμε στην παρούσα φάση. Πάντως υπάρχει μια κοινή δήλωση που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα διορθωτικό το ταχύτερο δυνατόν αυτή τη στιγμή έχει γίνει δεκτή η νομική βάση και αυτό θα κάνουμε. Και οι αρχές επί των δημοσιονομικών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν το αίτημα αυτό το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να μπορέσουμε πράγματι να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το επιπλέον Ταμείο Εγγύσεων. Τελειώνοντας να πω ότι εμείς σε επίπεδο ΝΤΕΦΚΟ είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής και σας ευχαριστώ για το σύνολο της εργασίας που κάνατε. Ο κύριος Πανιγκάλε, αν ακούσαμε καλά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με μας θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστούμε που μου δώσατε τη δυνατότητα σύντομα να αναφερθώ στα θέματα τα ανθρωπιστικά στον προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο. Να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο γενικότερα για τη στήριξή του στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαδικασίας. Γνωρίζουμε ότι η τελική έκβαση δεν ήταν η αναμενόμενη, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι είμαστε θα έλεγα συμβατοί με αυτά τα οποία προβλέπει το πολιετές δημοσιονομικό. Νομίζω λοιπόν ότι είχαμε ανάγκη 300 ή μάλλον έχουμε στη διάθεσή μας 300 εκατομμύρια για τις ε, μεταναστευτικές κρίσεις έχουμε κάποια άλλα επιπλέον κονδύλια για τις έκτακτες καταστάσεις αυτά έγινε πέρυσι, τα ίδια γίνονται και φέτος και είναι σχετικά συμβατά με αυτά τα οποία είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την πρόταση προϋπολογισμού του 2017. Βέβαια οι διαφορές παρέμειναν μεγάλες και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των διαφόρων αυτών. Τι ακριβώς θα κάνουμε. Καταρχάς έπρεπε να να καταρτήσουμε σωστά τις προτεραιότητές μας για την κατανομή των πιστώσεων στις διαφορετικές κρίσεις. Η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, βρισκόμαστε όμως στο τέλος. Έχουμε μια πρόταση απόφασης η οποία είναι υπό προετοιμασία. Έχουμε ένα συνολικό ποσό ε, για να το θέσουμε σε, ε, στα διαθέσιμα το οποίο είναι χαμηλότερο από ότι στο παρελθόν και δεν ξέρω αν καλύψει τις ανάγκες που έχουμε, που μπορεί να έχουμε σε σχέση με έκτακτες κρίσεις. Ο προϋπολογισμός για την ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να καλύψει επίσης και κάποιες πολιτικές αποφάσεις που πήραμε φέτος και τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε όπως σαν παράδειγμα τις αποφάσεις της διάσκεψης του Λονδίνου για τη Συρία και ταυτόχρονα τα ποσά τα οποία προβλέπεται να δοθούν στην Τουρκία για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. Όλα αυτά θα πρέπει να προσθεθούν στο σύνολο των ποσών που προβλέπονται για όλες τις άλλες κρίσεις. Είμαστε όμως πεπισμένοι ότι όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και το 2017 θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τα ποσά αυτά και στα πλαίσια του τμήματος 4 και στα πλαίσια της χρήσης του αποθεματικού για έκτακτες καταστάσεις το οποίο ελπίζουμε στα πλαίσια μιας ενδιάμεσης ε, αναθεώρησης ε, του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου να διευρύνουμε και στα πλαίσια των, ε, μέσων που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας και από άλλες πηγές όπως από εξωτερικά έσοδα εκτός προϋπολογισμού δηλαδή και τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν και για, τις χώρες μέλη και για τους πρόσφυγες και για άλλες μορφές συνεργασίας. Έχουμε λοιπόν να εργαστούμε με έναν περιορισμένο προϋπολογισμό, αυτό δεν είναι μυστικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας και να θυμίσω την προσπάθεια την οποία κάνουμε στις μεγάλες, στα πλαίσια της μεγάλης συνδιαλλαγής για το σύνολο της αποτελεσματικότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας και ταυτόχρονα να δούμε ακριβώς τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δωρήτριες χώρες και στην Ένωση. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Ντίβα για την ενημέρωσή σας. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερο χρήσιμη. Σας ευχαριστώ. Σύντομα όμως θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και το δικό μου προσωπικό για την εξαιρετική τους βοήθεια. Έχουμε λοιπόν καλύτερες ε, δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι περιμέναμε. Όχι αυτό που θα θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά ε, σας ευχαριστώ για την ενημέρωσή σας. Τώρα περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, το τελευταίο πριν πάμε στην κοινή συζήτηση με την ΑΦΕΤ. Πρόκειται για το Ταμείο για την Κολομβία. Τον Αύγουστο Ξέρετε ότι υπεγράφει μια ιστορική συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στα ΦΑΡΚ και την κυβέρνηση της Κολομβίας. Στο δημοψήφισμα στην Κολομβία δυστυχώς απερίφθη η πρόταση αυτή. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια νέα συμφωνία ανάμεσα στα ΦΑΡΚ και την κυβέρνηση που θα πάει την επόμενη εβδομάδα ε, προς έγκριση στο Κοινοβούλιο της χώρας και ε, σε λίγο καιρό θα θα δοθεί και το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη στον Σάντο, τον πρόεδρο της χώρας. Είναι χρήσιμο να έχουμε αυτή τη συζήτηση για να μάθουμε ακριβώς τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πώς ακριβώς θα δοθούν τα χρήματα αυτά. Ξέρουμε τι έγινε με το αντίστοιχο με το αντίστοιχο Ταμείο για την Αφρική και η κυρία Βιτσιένη θα μας δώσει πληροφορίες για το τι συμβαίνει και για το πώς μπορεί να εμπλακεί το Κοινοβούλιο και αν θα υπάρξει κοινοβουλευτικό έλεγχος επ' αυτού. Ευχαριστώ. Δεν θα σας κουράσω πολύ με τις λεπτομέρειες ε, και νομίζω πως ε, είναι καλή χρονική ε, ε, συγκυρία εδώ, γιατί μόλι τώρα ο συναδελφό έθεσε και το ερώτημα κατά πιστεματικά ταμεία αυτά τα trust funds. Όποιο λοιπόν έχει παρακολουθήσει τι ειδήσει κατά τι τελευταίε εβδομάδε, ε, σίγουρα θα είδε ε, την Κολομβία. Και γνωρίζετε, ή γνωρίζετε ότι μετά τη Συρία η Κολομβία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικά εκδιωγμένων ανθρώπων. Ε, δηλαδή ο πόλεμος, ο εμφύλιος ο πόλεμος εκεί λαμβάνει χώρα ε, εδώ και δύο γενιές ανθρώπων, εδώ και 50 χρόνια. Και αυτό βέβαια έχει πολύ ε, σημαντικό αντίκτυπο και στις γειτονικές χώρες, ειδικότερα το Εκουαδόρ. Η ε, περιπλοκότητα των ενευτικών διαδικασιών ήδη αναφέρθηκε, η συμφωνία με το ΦΑΡΚ, δηλαδή το Κογκρέσο σήμερα ξεκινάει τη συζήτηση της νέας ενευτικής συμφωνίας, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες εάν δεν κινηθούμε γρήγορα με την ενευτική διαδικασία θα καταλάβουν ταχύτατα το κενό ε, που αφήνει σε αυτό το πολύ περίπτωκο πλαίσιο ε, το ΦΑΡΚ. Οπότε χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να σας αναφέρω ε, κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό το Trust Fund και πραγματικά δεν θα πρέπει να το θεωρήσετε ίδιο με τα υπόλοιπα. Είναι ένα σχετικά μικρό Trust Fund σε σχέση με τα υπόλοιπα, το οποίο όμως μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Ε, όχι μόνο υποστηρίζει ε, την ε, ειρηνευτική συμφωνία και η οποία αναμένεται στις 12 Δεκεμβρίου να συζητηθεί για να λάβει και, σε σχέση με το βραβείο Νομπληρής που έλαβε ο κύριος Σάντος. Θα τον αποδεχτούμε λοιπόν εδώ. Και έτσι λοιπόν δύο εβδομάδες ε, μα ε, απομένουν ε, για την υιοθέτηση αυτού του Trust Θέλουμε λοιπόν να καταδείξουμε ότι με αυτό το ταμείο έχουμε επιλέξει το καλύτερο εργαλείο για να υποστηρίξουμε την ευθυκή διαδικασία στην Κολομβία και πραγματικά είναι κατάλληλη χρονική συγκυρία. Αν συγκρίνουμε αυτό το ταμείο με τα υπόλοιπα θα δούμε ότι έχει το μεγαλύτερο αριθμό χορηγών. Έχει δηλαδή ήδη από την δημιουργία του 14 κάτι μέλη που συμμετέχουν. Άλλα ε, trust fund ξεκίνησα με λίγες ε, χώρες και μετά σιγά σιγά αυξήθηκαν οι χώρε χορηγοί. Αντιθέτω, αυτό το ταμείο ξεκινάει με, πολλές, ε, με πολλά κράτη-μέλη και ελπίζω ότι θα προσθεθούν κι άλλα. Υπάρχουν άλλα έξι κράτη-μέλη τα οποία αναλογίζονται τη συμμετοχή του σε αυτό το ταμείο. Ε, δεν είμαστε εμεί οι οποίοι είχαμε αυτή την ιδέα. Η κολομβιανή κυβέρνηση ήταν εκείνη η οποία απευθύνθηκε σε εμά και μα ε, ε, ζήτησε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργαλείο και πραγματικά ε, βρήκανε βίκο αότα ε, από τη, και από την πλευρά των κρατών μελών, για παράδειγμα και στο πλαίσιο της περσινής συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΑΚ. Εκεί δηλαδή συμφωνήθηκε αυτή η ιδέα, γιατί υπήρχαν και υψηλή αξιωματούχοι εκεί, για παράδειγμα και ο υπουργό Εξωτερικών από το Μεξικό, ο οποίο ανέφερε ακριβώ στην ομιλία του εδώ ότι πραγματικά δεν θα πρέπει να υποτιμήσετε ω Ευρωπαϊκή Ένωση τον ρόλο που μπορείτε να παίξετε στην περιοχή περιοχή τη Λατινική Αμερική και σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία μέσω ακριβώ ενό ε, τέτοιου ταμείου. Τι είναι σημαντικό σε σχέση με αυτό το ταμείο. Εντάσσεται σε αυτό το νέο όραμα τη ε, ειρηνευτική ε, πολιτική, σε αυτή την κοινή αντίληψη την οποία συζητάτε. Δηλαδή τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε μια κοινή συντονισμένη δράση και κατά συνέπεια έχουν και πολύ μεγαλύτερο μοχλό σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπό του. Δηλαδή μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο αυτό η ε, ε, κολομβιανή κυβέρνηση έχει αναλάβει τις δικές της ε, ευθύνες εδώ και μας είπε ότι από νωρίς ότι θέλουμε τις δικές σας δικές σας εμπειρογνωμοσύνη, θέλουμε το δικό σας soft power, θέλουμε δηλαδή τα όσα έχετε επιτύχει σε εσά να προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε και εμείς για να τα επιτύχουμε. Και προφανώ δεν θα έχουν επιληθεί όλα τα ζητήματα και η Γενική θα πρέπει να συνεχίσει τι εργασίε που κάνει σε αυτή την ε, περιοχή, γιατί υπάρχουν και ε, ένα σωρό περιοχέ στι οποίε δεν έχουμε πρόσβαση ακόμα. Ε, και όταν είχαμε συζητήσει με κάποιου προσώπου και δήμων και κοινοτήτων, δημάρχου και άλλου που είχαν έρθει στην Μποκοτά για να συζητήσουμε τα ζητήματα, μου έκαναν, προσκάλεσαν ε, να τους επισκεφθώ ε, στους Δήμους και στις κοινότητες τους και τους είπαν ναι, ε, φυσικά αστειευόμενο ότι να έρθω να σε επισκεφθώ, αλλά πώς θα γυρίσω πίσω στην Πόγκοτα και ε, συμφώνησαν μαζί μου. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια εργαστήρια εντό εισαγωγικών για την ερευνητική διαδικασία που εξετάζουν ακριβώ το πόσο μπορούν να δημιουργηθούν οικονομικέ δυνατότητε και δυνατότητε διαλόγου για αυτέ τι κοινότητε. Δεν θέλω να αναφερθώ βέβαια σε όλε τι ομότητε και όλα τα, τα βία γεγονότα που έχουν λάβει η χώρα σε αυτέ τι ε, περιοχέ, αλλά πραγματικά μέσω ακριβώ τη δημιουργία αυτών των ειρηνευτικών εργαστηρίων και μέσω των προσπαθειών που έχουμε κάνει, έχουμε επιτύχει την ε, ε, τέτοιε περιοχέ. Άρα λοιπόν έχουμε δείξει ότι στην Κολομβιανή κυβέρνηση ότι αν θέλει η ειρηνευτική διαδικασία διαδικασία αναστευτεί με επιτυχία, θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει και τη δική μας ε, ε, δύναμη. Δηλαδή η Ευρώπη δεν έχει οικοδομηθεί μόνο μέσω της Για παράδειγμα, τα παραδείγματα στην Ιρλανδία μας δείχνουν το τι κάνουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε και τον εκπρόσωπο από την Ελλάδα που συμμετέχει. Και ο τις επιτροπές από την πλευρά του Φάρκο το όνομα Μοσέκου, ε, αναγνώρισε ακριβώς το ρόλο που μπορεί να παίξει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβόλιο τώρα μας ζήτησε να ε, ε, τευθεί, να, να μπει το Ταμείο και μέσα στο γενικότερο πρόγραμμα της ανάπτυξη τη υπέδρου, Γιατί βέβαια από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα του, ότι υπήρχε δηλαδή πλήρη απουσία του κράτου και των δημοσίων υπηρεσιών, κανένα έλεγχο και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν ε, ακριβώς εκεί μας ζητήθηκε να παρέμβουμε, αλλά βέβαια είναι και ο πιο δύσκολος ε, τομέας για παρέμβαση. Ε, αυτό όμως μας ζητήθηκε και φυσικά εδώ χρειάζεται να δημιουργηθεί και περισσότερη εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, γιατί είναι φοβισμένοι δηλαδή οι πολίτες σε αυτές τις υπαίθριες περιοχές δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε ε, σε αυτούς τους ανθρώπους την εντύπωση ε, που έχουν για παράδειγμα ε, οι κάτοικοι στην Ήπεθρο της Βενεζουέλας ως προς τους τσαβίστας. Δηλαδή θέλουμε πραγματικά να τους δείξουμε ότι είμαστε εκεί και να τους βοηθήσουμε. Θέλουμε λοιπόν γενικά να ενισχύσουμε το ρόλο που παίζει το κράτος, να καταπολεμήσουμε τη βία και πραγματικά θεωρούμε ότι μπορούμε να δώσουμε εδώ προστεμένη αξία από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών. Οι προτεραιότητε είναι λοιπόν η υποστήριξη τη αγροτική πολιτική και η αναζωογόνηση τη αγροτική παραγωγή και βιωσιμότητα και η συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Όλα αυτά βέβαια θα συνοδευτούν από τεχνική υποστήριξη και από εμπειρογνωμοσύνη των συμμετοχών των κρατών μελών. Ε, είναι λοιπόν φιλόδοξα αυτά τα όσα θέλουμε να επιτύχουμε. Ε, και ε, βέβαια είναι και το ζήτημα του κόστους. Αλλά είναι πραγματικά φτηνό το εισαγωγικό αυτό το ταμείο. 70 εκατομμύρια ε, ευρώ θα κοστίσει στον προπολογισμό της Ένωσης. Είμαστε πολύ ε, περήφανοι γιατί συμμετέχει και ακόμα 2 εκατομμύρια και 22 εκατομμύρια βουλευτά των κρατών μελών, δηλαδή στο σύνολό του 95 εκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευθεί για αυτό το Trust Fund και πραγματικά είμαστε ένας σημαντικός εταίρος. Η Κολομβία βέβαια έχει υπολογίσει πως ε, η ειρηνευτική διαδικασία θα κοστίσει στον γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε τώρα ε, τα 100 εκατομμύρια ευρώ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής ε, δεν θα καλύψω μεγάλο τμήμα αυτών των κονδυλίων, αλλά πραγματικά έχουν έχει τεράστιο αντίκτυπο αυτή η υποστήριξη γιατί δίνουμε αυτό το μήνυμα της υποστήριξης και της ανάληψης της δέσμευσης απέναντι σε αυτή την ενευτική διαδικασία. Ότι δηλαδή όχι μόνο υποστηρίζουμε στα λόγια την ενευτική διαδικασία αλλά ε, προβαίνουμε και σε πράξεις. Οπότε ε, αυτό που θα κερδίσουμε με αυτή την υποστήριξη με τα 100 εκατομμύρια ευρώ θα είναι πολύ περισσότερο ε, και βέβαια θα υπάρξει και ταυτόχρονα χρηματοδότηση από τους του Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομή και θα εργαστούμε μέσω μηχανισμών παροχής της βοήθειας. Δηλαδή, θα ε, παράσχουμε αυτή τις ενισχύσεις και μέσω των δικών μας μηχανισμών, όχι άλλων διεθνών οργανισμών. Ε, και αυτό είναι και σημαντικό ως πως το, για παράδειγμα, πού θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας, θα περιοριστούμε σε συγκεκριμένες ε, περιφέρειες, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές όπου ήδη έχουμε εργαστεί. Και ε, Τέλο να σα πω ότι το καινοτόμο στοιχείο αυτού του ε, Trust Fund είναι ότι θα εδρεύει στην ε, Μποκοτά. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα Trust Funds έχουν την έδρα του στι Βρυξέλλε, ενώ το συγκεκριμένο θα έχει την έδρα του στην Μποκοτά. Στι 12 Δεκεμβρίου θα υπογραφεί λοιπόν αυτό το Trust Fund και θα λειτουργήσει όπω όλα τα υπόλοιπα. Και κάθε, οποτεδήποτε το, το Κοινοβούλιο ε, μας ζητήσει περισσότερη ενημέρωση, είμαστε στη διάθεση να το ενημερώσουμε. Ε, Τησίως ούτω ή άλλω θα γίνεται μια ένας απολογισμός εδώ στο Κοινοβούλιο και αναμένουμε ότι το ε, Ταμείο θα τεθεί σε λειτουργία, θα αρχίσει να ε, λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2017. Ευχαριστώ πολύ, λέει, η Πρόεδρος, ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και αναμένουμε ε, με ενδιαφέρον την έρευνση τη χρηματοδότηση. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι έχουν να θέσουν ερωτήματα. Ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Κανονικά τα trust fund δημιουργούνται για να επιταχύνουν τις ε, ε, δόσεις. Ε, έχουμε διάφορους δωρητές οι οποίοι έρχονται για να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Πώς λοιπόν θα διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα του συγκεκριμένου Trust Fund θα ελέγχονται ώστε να χρησιμοποιούνται για τα ε, προγράμματα τα οποία είναι αναγκαία όπως είναι για παράδειγμα έχουμε την ε, Χαϊτή η οποία παραμένει ε, σε χαοτική κατάσταση Πώς θα γίνεται ακριβώς λοιπόν ο έλεγχος Έχουμε σήμερα δορυφόρους, οπότε μπορούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται ε, στις διάφορες τοποθεσίες. Θα χρησιμοποιήσετε δορυφόρους που δορυφόροι οι οποίοι μπορούν να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα σημεία για να ελέγξουν το ε, τι θα συμβεί. Ποιος λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, θα ελέγχετε τι γίνεται. 100 σχολεία χτίστηκαν, 200 πηγάδια άνοιξαν. Τι ακριβώς θα κάνετε άλλος ε, συνάδελφος που θέλει να θέσει ε, ένα γρήγορο ερώτημα. Διότι ε, δεν έχουμε χρόνο. Εγώ προσωπικά έχω μια καλή εικόνα του συγκεκριμένου ε, Trust Fund. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η IT είναι επίσης ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί. Υπάρχουν δύο θέματα όμως. Ναι, το Transplant είναι κάτι πολύ πιο ευέλικτο και έχει ε, τέσσερις φορές μεγαλύτερη ταχύτητα. Όμως εδώ μιλάμε για λιγότερο από 100 εκατομμύρια ε, όταν εσείς ε, ασχολείστε με δράσεις ε, στην Αφρική μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα ποσά. Εμείς θα κάνουμε μικρές δράσεις που όμως έχουν μεγάλο αντίκτυπο από άποψης πολιτικής και ανάπτυξης. Είναι δράσεις που θα επικεντρώνονται στα όσα έχουμε συζητήσει. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε δορυφόρους. Ρώτησα για drones και αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά για τοποθεσίες για παράδειγμα ε, που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ε, έρευνα ε, δεν κάνουμε τίποτα, αυτό είναι ο κανένα, αν δεν έχουμε επισκεφθεί την τοποθεσία. Θέλουμε να ξέρουμε ποιο θα λάβει στο τέλο τα χρήματα, πηγαίνουμε, ελέγχουμε στην Αιτία αποδείχθηκε όπου ε, δυσκολευόμασταν να επισκεφθούμε κάποιες, κάποιες περιοχές. Εκεί αποτύχαμε. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Κάτι ακόμα για την Κολομβία. Ίσως να μην το θυμάστε επειδή ασχολείστε με πολλά και η Λατινική Αμερική δεν αποτελεί προτεραιότητά σας έχουμε υποστηρίξει ότι η Κολομβία είναι μια ιδιαίτερη περίστοση ε, και επενδύουμε μονάχα 270 εκατομμύρια οπότε ε, όσον αφορά την ε, συμφωνία ειρήνης θα βρισκόμασταν σε άσχημη κατάσταση εάν δεν ε, ασχολούμασταν με αυτό και, αυτό και γι' αυτό αποφασίσαμε ότι η επένδυσή μας θα πρέπει να φτάσει εκεί. Το ίδιο ισχύει ε, και για, το, για τον Ισημερινό διότι τα όσα συμβαίνουν ε, στην Κολομβία έχουν συνέπειες ε, όπως είναι για παράδειγμα η πεντανάστευση και οι εγκληματικές δραστηριότητες και σε γειτονικέ ε, χώρες. Το 2017 λοιπόν θα επικεντρωθούμε στην Κολομβία. Σίγουρα όμως θα σας δείξουμε φωτογραφίες. Ναι, θέλουμε να ε, συνεχίσουμε να λαμβάνουμε ενημέρωση για το συγκεκριμένο Trans Fund, διότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα και εν τέλει αφορά τη ζωή ανθρώπων, άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν αξιοπρεπείς ε, συνθήκες διαβίωσης. Συνάδελφοι, τώρα έχουμε την κοινή συνάντηση ε, με την ΑΦΕΤ για τη Συρία και όσοι δεν είσαστε εδώ από ό,τι φαίνεται το Χαλέπι έχει πέσει οπότε θα υπάρχει μια σοβαρή ανθρωπιστική ε, κατάσταση εκεί πέρα ε, σε 5 λεπτά στην αίθουσα 2Q2. Σας ευχαριστώ.